Λοιπόν, παραδοσιακά ε, με βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων της χώρας που έχει την Προεδρία του Συμβουλίου κάθε φορά. Καλώς ορίζω και πάλι τον κύριο Σταμενίτη, καλώς ορίσατε στην Επιτροπή μας και θέλω να σας πω ότι τα μέλη της Επιτροπής μας περιμένουν να ακούσουν αυτά που έχετε να μας πείτε για τις προτεραιότητες, τις προκλήσεις και ό,τι έχει να αντιμετωπίσει η Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου. Επίσης, θα θέλαμε να ακούσουμε και θέματα ευρωπαϊκά, αλλά και εκείνα που άπτονται της μεταρρύθμισης κοινή αγροτικής πολιτικής. Μετά την παρουσίασή σας θα έχουμε χρόνο για συζήτηση και ερωτήσεις. Παρακαλώ, έχετε μέσα στο λόγο, κύριε Σταμενίτη. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι μέλη της Επιτροπής, βρίσκομαι σήμερα μαζί σας με σκοπό να σας παρουσιάσω την πραγματικότητα της ελληνικής γεωργίας τις απόψεις του Ελληνικού Κοινοβουλίου σχετικά με την αναθεώρηση της κοινή γεωργικής πολιτικής, αλλά και τις στοχεύσεις ελληνικής πλευράς από την εφαρμογή της. Κυρίες και κύριοι, εσείς εδώ και δύο χρόνια εργάζεστε για τη νέα κοινή γεωργική πολιτική που περιλαμβάνει τέσσερις βασικούς κανονισμούς. Τον πρώτον τις άμεσες ενισχύσεις, το δεύτερο την ενιαία κοινή οργάνωση αγοράς των γεωργικών προϊόντων, την τρίτη την αγροτική ανάπτυξη, και την τέταρτη τον οριζόντιο κανονισμό για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και τον έλεγχο της κοινή γεωργικής πολιτικής. Ήδη υπάρχουν μεταβατικές ρυθμίσεις για το 2014, ενώ από 1η 2015 θα έχουμε πλήρη εφαρμογή του νέου καθεστώτος. Από ελληνική πλευρά η εμπειρία της εφαρμογής της προηγούμενης περίοδου μας έχει διδάξει πολλά και η υιοθέτηση της νέας μας δίνει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα προγραμματίσουμε και θα ιεραρχήσουμε τους στόχους που θέτουμε για την ελληνική γεωργία δηλαδή να καταφέρουμε βήμα-βήμα με βασικό εργαλείο τη νέα κοινή γεωργική πολιτική να επιτύχουμε όσα ορεματιζόμαστε για την ελληνική γεωργία μέχρι το 2020. Και για να φτάσει μια πολιτική στο αποτέλεσμα που επιθυμεί η πολιτεία και η κοινωνία πρέπει να υπάρχουν οι βασικοί σταθμοί που ουσιαστικά θα υποδείξουν τον δρόμο και τις επιλογές. Από την πλευρά μας υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι. Συγκεκριμένα. Πρώτον, μια ελληνική γεωργία ανταγωνιστική προσανατολισμένη στην παραγωγή μέσω της μεταπητικής βιομηχανίας ποιοτικών τροφίμων υψηλής προ... προστατευμένης αξίας, ώστε να διαδραματίσει το ρόλο που της αναλογεί στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Δεύτερον, μια ελληνική γεωργία ικανή να ανταποκριθεί στο σκοπό της, δηλαδή στην εξασφάλιση της επιστηστικής ασφάλειας και της δημόσιας υγείας. Τρίτον, μια ελληνική γεωργία εξωστρεφής, ώστε να συμβάλλει στην ενδυνάμωση των εξαγωγών μας, και στη βελτίωση του εμπορικού συζωγίου της χώρας μας. Τέταρτον, μια ελληνική γεωργία ικανή να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή και τις νέες προκλήσεις που παρουσιάζονται. Και πέμπτον, τελευταίο, όχι λιγότερο σημαντικό, η ενδυνάμωση των συνεργειών στην ελληνική περιφέρεια, ώστε να προβάλλουμε το πολιτιστικό, περιβαντολογικό, γαστρονομικό και τουριστικό πλούτο της χώρας μας ως βασικό εργαλείο περιφερειακής ανάπτυξης να εξασφαλίσουμε έτσι ένα βιωτικό επίπεδο του αγροτικού μας πληθυσμού. Σε μια χώρα σαν την Ελλάδα που περίπου το 40% του πληθυσμού κατοικεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η ανάπτυξη της περιφέρειας αποτελεί τη μεγάλη μας πρόκληση. Για να προχωρήσουμε όμως στην υλοποίηση των στόχων, θα πρέπει να πρώτα να δούμε και να αναλύσουμε τι συμβαίνει σήμερα, ποια είναι η υπάρχουσα κατάσταση, τι συμβαίνει σήμερα στην ελληνική γεωργία. Ο ελληνικός αγροτικός τομέας χαρακτηρίζεται από περιορισμένη ανταγωνιστικότητα που απορρέει από κοινωνική δομή και τις διαρθωτικές και φυσικές ανισότητες μεταξύ των διαφόρων γεωργικών περιοχών της χώρας. Η Ελλάδα είναι μια χώρα ορεινή με πλούσιο οριζόντιο εδαφικό διαμελισμό και έντονο ανάγκληφο αποτελούμενη από δύο περιοχές, την υπηρετική και την ισιωτική. Το βορειοδυτικό τμήμα της χώρας δέχεται τις περισσότερες βροχοπτώσεις γι' αυτό και χαρακτηρίζεται από κλίμα υγρό μεσογειακό, σε αντίθεση με το νότιο-ανατολικό τμήμα που χαρακτηρίζεται από ξηρό μεσογειακό. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ο βοροδυτικό τμήμα της χώρας χαρακτηρίζεται από πλεόνασμα υδατικού ισοζυγίου, ικανό να συντηρήσει μια πιο δυναμική γεωργική παραγωγή, όμως στα λιγοστά παιδινά τμήματα σε αντίθεση με τον νότιο ανατολικό που παρουσιάζει έλλειμμα και συνεπώς μικρότερη ικανότητα γεωργικής παραγωγής. Δεν είναι δε τυχαίο ότι σε αυτό το τμήμα αναπτύχθηκε αρχικά ο τουρισμός. Από την άλλη μεριά, η παραλλακτικότητα μορφολογίας και κλίματος σε μια τόσο περιορισμένη έκταση συντηρεί μια μοναδική βιοπικιλότητα που απαριθμεί ποικίλα ενδυμικά είδη και την οποία έχουμε χρέος να προστατεύσουμε και να αναπαράγουμε ο ιδιαίτερος χαρακτήρας ελληνικής γεωργίας, ας μου επιτραπεί η έκφραση, η μοναδικότητα της ελληνικής γεωργίας τηρουμένου των αναγιών, αναδεικνύεται και μέσα από την πληθώρα των προβλημάτων που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και τα οποία στοχεύουμε να ελαχιστοποιήσουμε μέσα στο πλαίσιο των κοινών ευρωπαϊκών πολιτικών. Είναι κοινό τόπο σήμερα ότι η εφαρμογή μια πολιτικής σχεδιασμένη για όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης δημιουργεί ορισμένα προβλήματα. Και αυτό συμβαίνει όχι επειδή δεν είναι σωστός ο σχεδιασμός, αλλά λόγω του ότι έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα η γεωργική δραστηριότητα. Και ίσως αυτός είναι ο λόγος που βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ορισμένα διλήμματα, όπως αυτό της διαφοροποίησης του νέου δικαιώματος τόσο μεταξύ των κρατών μελών, όσο και εντός των περιεχών ενός κράτους μέλους. Συνεπώς, χαιρετίζουμε την προσπάθεια για θεσμοθέτηση ενός πιο ευέλικτου και αποτελεσματικού πλαισίου για τις άμεσες ενισχύσεις στο γεωργικό τομέα που οδηγεί στην σταδιακή σύγκληση των ενισχύσεων ενός πλαισίου πιο πράσινου αλλά συγχρόνως και πιο δίκαιο για τους παραγωγούς. Για την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επεξεργάζεται τέσσερα διαφορετικά σενάρια και τα οποία σας αναφέρω επιγραμματικά. Το πρώτο προβλέπει την χώρα ως μία ενιαία περιφέρεια. Το δεύτερο χωρίζει τη χώρα σε 13 διοικητικές περιφέρειες. Το τρίτο χωρίζει τη χώρα σε δύο περιφέρειες, πρώτη των καλλιεργούμενων εκτάσεων και δεύτερη των βοσκοτόπων. Και το τέταρτο περιλαμβάνει τέσσερις περιφέρειες, πρώτη καλλιεργούμενες πεδινές, δεύτερη καλλιεργούμενες ορεινές εκτάσεις, τρίτη βοσκότοπη παιδινών και τέταρτη ορεινών εκτάσεων αντίστοιχα. Ανεξάρτητα την επιλογή του σενάριου, η Ελλάδα εξασφαλίζει του βασικού στόχου που τίθενται με την εφαρμογή της νέα κοινή γεωργική πολιτική, δηλαδή την εξισορρόπηση της μοναδιαία αξίας δικαιώματο ανάμεσα στι διοικητικέ περιφέρειε, καθώς και ανάμεσα στου παραγωγού. Παράλληλα, επιτυχάνει τη μετακίνηση χρημάτων μεταξύ των παραγωγών. Εκτιμάται ότι οι κερδισμένοι θα είναι περισσότεροι των χαμένων. Στόχος του Υπουργείου και της χώρας μας είναι επιλογή εκείνου του σενάριου που μεγιστοποιεί τα ωφέλη της νέας κοινή γεωργικής πολιτικής για τη χώρα μας και συγκεκριμένα. Πρώτον, στην ενίσχυση της αηφορίας του γεωργικού χώρου μέσω των άμεσων ενισχύσεων, κυρίω λόγος του μέτρου παρασυνίσματος και της ενσωμάτωσης στην πολλαπλή συμμόρφωση της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά και της οδηγίας για την αηφόρο χρήση των φυτοπαρμάκων που σε συνδυασμό με τα σύγχρονα εμπορικά πρότυπα θα μειώσουν τις ροές. Δεύτερον, στη βελτίωση της επάρκειας των προϊόντων, αφού θέτουμε ως στόχο τον περιορισμό των εκτάσεων σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 10% του συνόλου των εκτάσεών μας. Και αυτό θέλουμε να το πετύχουμε τη δυνατότητα που παρέχεται στο κράτο μέλος να ορίσει ελάχιστη γεωργική δραστηριότητα στις εκτάσεις προκειμένου να απολαμβάνουν τις ενισχύσεις που τους αναλογούν. Τρίτον, στην περαιτέρω προώθηση της διαφοροποίησης των νέων παραγόμενων προϊόντων, η οποία με τη νέα κοινή γεωργική πολιτική είναι δεδομένη, καθώς η συνέχιση του καθεστώτος της αποσύνδεσης των ενισχύσεων θα αναγκάσει τους γεωργούς να παράγουν όλο ένα και περισσότερο για την αγορά και να ανταποκρίνονται στη ζήτηση. Τέταρτον, συγχρόνως η παραγωγή κινήτρων που μας προσφέρει η νέα πολιτική με τη μορφή συνδεμένων ενισχύσεων θα μας επιτρέψει την αναδιάρθρωση της παραγωγής προς εκείνους τους τομείς για τους οποίους παρουσιάζεται σημαντική υστέρηση ώστε να βελτιώσουμε το εμπορικό συζύγιο της χώρας. Πέμπτον, προσανατολιζόμαστε στην ενίσχυση των ζωοτροφών ώστε να μειώσουμε το κόστος παραγωγής των ζωοκομικών προϊόντων μας αφού η φέτα και το γιαούρτι είναι ο σημαντικότερος πρεσβευτής της ελληνικής γεωργίας. Έκτον, στην ανανέωση του γεωργικού πληθυσμού στοχεύουμε σε εισαγωγή τουλάχιστον 8.000 νέων γεωργών αρχηγών εκμεταλλεύσεων στο γεωργικό τομέα. Έβδομον, στην ορθή διαχείριση των υδάτων με τη μείωση της κατανάλωσης αρδευτικού νερού και την αποφυγή της ρήπανσης. Όγδο, στην ανάδειξη της ποιότητας των προϊόντων μας ως συγκριτικού πλεονεκτήματος έναντι των άλλων χωρών, η οποία σε συνδυασμό με τη σχεδιαζόμενη εξωστρέφεια του αγροτικού τομέα κρίνουμε ότι θα επιφέρει αθρηστική αύξηση της προστιθέμενης αξίας της γεωργίας περισσότερο από 15%. Και ένατον, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η κοινή αγροτική πολιτική διαθέτει στο δεύτερο πυλώνα της μέσω της αγροτικής ανάπτυξης πλειάδα πιθανών μέτρων τα οποία μπορούν να ενεργοποιηθούν και να αποφέρουν σημαντικά ωφέλη στο γεωργικό τομέα και ο στόχος των πολιτικών μας είναι η άβληση και η θεραπεία των επιπτώσεων που έχει το συγκεκριμένο φαινόμενο. Κυρίε και κύριοι, θα ήθελα, κλείνοντα την εισήγησή μου, να σταθώ σε ορισμένα ζητήματα που ανέφερε ο Πρωθυπουργό τη Ελλάδα και Προεδρεύων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, κ. Αντώνη Σαμαρά, στην ομιλία του, τα οποία θα απασχολήσουν την Ευρώπη στα επόμενα χρόνια. Πρώτον, η τόνωση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνοχής, το ένα προϋπόθεση του άλλου που μπορούν να συμβαδίσουν αρμονικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία. Δεύτερον, η στήριξη του κοινού νομίσματος και η ενίσχυση της Εμπιστοσύνη της κοινωνίας και των πολιτών στην ευρωπαϊκή ιδέα. Τρίτον, η λύση στο μεταναστευτικό πρόβλημα μέσω της ομικής διαχείρισης από την Ένωση. Και τέταρτον, η όθηση και η νέα πνοή στις θαλάσσιες πολιτικές της Ένωσης έκρινε απαραίτητη αυτή τη φαινομενικά εκτός πλαισίου αναφορά, γιατί για εμάς η οικονομική κρίση παρά τις δυσκολίες που μας επέφερε, μας έμαθε ότι οι πολιτικές επιλογές μέσα σε μια πολιτική και οικονομική ένωση δεν έχουν αξία όταν ασκούνται μονομερώς. Ότι οι λύσεις δεν δίνονται μονόπλευρα και το πρόβλημα δεν είναι ατομικό. Η Ελλάδα βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού, όμως με σοβαρότητα και ορθολογικές επιλογές κατάφερε να ξεπεράσει τον κίνδυνο, αποφεύγοντα τι εύκολε λύσει αγνοώντας φωνές λαϊκισμού και καταστραφολογίας μέσω και έξω από τη χώρα και χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία που μας παρέχει η δημοκρατία, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε την παραμονή μας στην οικονομική ζώνη του ευρώ, να σταθεροποιήσουμε την οικονομία μας και να πετύχουμε πρωτογενές πλεόνασμα περισσότερο από αυτό που είχε προβλεφτεί, από όσο υπολογίζαμε. Με την προσπάθεια να συνεχίσετε με την προώθηση όλων των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων για τη μείωση γραφειοκρατίας, δημιουργούμε ένα περιβάλλον σταθερό και ασφαλέ για τι ιδιωτικέ επενδύσει που θα μα βοηθήσουν στον αγώνα που δίνουμε για την τόνωση τη ανάπτυξη, τη μείωση ενεργεία και την ανίσχυση του γεωργικού τομέα. Και τέλο, ενισχύοντα το ρόλο τη δικαιοσύνη, αντιμετωπίζουμε σοβαρά και με αποτέλεσμα τη διαφθορά, ένα φαινόμενο που κόσσε τόσο οικονομικά όσο και την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματο. Με σταθερά βήματα και αποφασιστικότητα η Ελλάδα διορθώνει όλα τα αίτια που την οδήγησε στην οικονομική κρίση αλλά και τα λάθη του προγράμματο που είχε συμφωνηθεί με του εταίρου. Κυρίε και κύριοι, το παράδειγμα τη σημερινή Ελλάδα που στάθηκε στα πόδια τη και τα καταφέρει μέρα με τη μέρα περισσότερο, μα δείχνει τον δρόμο για περισσότερη Ευρώπη, για κοινέ πολιτικέ και συλλογική δράση. Θα κλείσω χρησιμοποιώντα τα λόγια του Πρωθυπουργού στην ομιλία που έδωσε την περασμένη Πέμπτη στην συνάντηση τη Αθήνα με θέμα τολμήστε τη δημοκρατία στα πλαίσια τη ελληνική προεδρία. Είπε, ο καθένας μόνος του, είτε πρόκειται για μεγάλο κράτος, είτε πρόκειται για μικρό κράτος, θα κερδίσει πολύ λιγότερα από ό,τι μπορούμε να κερδίσουμε όλοι μαζί. Και ο καθένας μας θα κινδυνεύσει πολλά περισσότερο αν μείνει μόνος του, ενώ όλοι μαζί θα είμαστε πιο δυνατοί και πιο θωρακισμένοι. Το ίδιο πιστεύουμε για την εφαρμογή της νέας κοινή γεωργικής πολιτικής, γιατί τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικό τομέα σε ολόκληρη την Ευρώπη, όπω για παράδειγμα η κλιματική αλλαγή, το υψηλό κόστο παραγωγή, είναι κοινά. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας και την πρόσκληση και την ευκαιρία που μας δώσατε να εκθέσουμε τις απόψεις του Ελληνικού Κοινοβουλίου στην Επιτροπή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στα μέλη της Επιτροπής μας. Η κυρία Γκαρσία έχει το λόγο και μετά ο κύριος Άγνιο. Πρώτα η κυρία Γκαρσία λοιπόν. Κυρία Γκαρσία έχετε το λόγο. Ξέρετε Εμένα με λένε Εράντς Γκαρσία. Υπάρχει και άλλη Γκαρσία, η κυρία Εράτσε Γκαρσία. Οπότε μπερδεύτηκα. Εγώ λέγομαι Εράντς Γκαρσία. Ε, ευχαριστώ, εν πάση περιπτώσει. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της Βουλής των Ελλήνων, τον κύριο Σταμενίτη, τον κύριο Βουλευτή, γιατί μας είπε ποια είναι η ελληνική γεωργία και ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Τα γνωρίζουμε αυτά γιατί ο συνάδελφος Γιώργος Παπαστάμκος που αποσιάζει εδώ και λίγο καιρό μας ενημέρωνε για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Και θέλω να ευχηθώ επευκαιρία περαστικά στον κύριο Παπαστάμκο το συντομότερο. Σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή και με χαρά πρέπει να σας πω. Πολύ καλά μιλήσατε για τον τρόπο στον οποίο ε, ε, κατανέμεται ο πληθυσμός, ότι είναι πολύ ε, μεγάλες οι δύο μεγάλες πόλεις και η ύπεθρος που σε γενικές γραμμές είναι αραιοκίνητη κατοικημένη. Ακριβώς η Γεωργία αυτό το καθήκον έχει και η κτηνοτροφία να κρατάει τον κόσμο στην ύπεθρο και θα πρέπει η Γεωργία και η κτηνοτροφία να είναι τρόπος ε, που να μπορεί ο κόσμος να κερδίζει τη ζωή του και ε, να ζει από αυτή σε όλη την επικράτεια. Και στη συνέχεια έρχεται η βιομηχανία τροφίμων για τα γεωργικά και τα δασοκομικά προϊόντα. Είναι πολύ βασική ε, κινητήρια δύναμη ε, μαζί με τα προϊόντα με ονομασία προέλευσης, γεωγραφικούς προδιορισμούς, παραδοσιακές ε, πρακτικές και σπεσιαλιτέ κτλ. Θα ήθελα να αναφερθώ επίσης σε ένα σημείο που μιλήσατε για την κοινή γεωργική πολιτική και τις ενισχύσεις. Προσπαθήσαμε και νομίζω ότι καταφέραμε να τους συμφωνήσουμε στην ΚΑΠ να υπάρχουν ε, διακοιμάνσεις όσο γίνεται πιο ισόρροπες και πιο δίκαιες στις ενισχύσεις που λαμβάνουν οι παραγωγοί και στην κατανομή, σε αυτόν τον καταμερισμό προς τη συνοχή μεταξύ κρατών και μεταξύ παραγωγών θα πρέπει να υπάρχουν όσο γίνεται λιγότερες απώλειες και ζημιές για τους παραγωγούς. Ελπίζω σε όλα τα κράτη-μέλη τώρα η εφαρμογή της ΚΑΠ θα διατηρήσει αυτό το πνεύμα που ξεκίνησε από εδώ, δηλαδή ότι πηγαίνουμε προς ε, μία ισότητα στην Ευρώπη μεταξύ των παραγωγών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκε που είναι δυσμενεί και πολύ σκληρέ σε ορισμένα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σα, σα ευχαριστώ για την παρουσία σα και που μα ε, εξηγήσατε λίγο παραπάνω πώς έχει πραγματική γεωργία στα κράτη-μέλη και θα σας ήμουν ευγνώμων αν μπορούσατε να μας πείτε ε, πώς βλέπετε το πακέτο για την προώθηση που αυτό τον καιρό διαπραγματεύονται, ε, πώς φαντάζεστε εκεί τις εξελίξεις και την πορεία του. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κύριος Άγνιου και μετά ο κύριος Ντές. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Ακούσαμε τις απόψεις σας για το τι συμβαίνει, όπως ξέρετε, φαντάζομαι, γνωρίζετε. Οι ευρωβουλευτές εδώ στην Επιτροπή Γεωργίας δεν ε, είναι καθόλου ικανοποιημένη από τις ε, καταξιδότηση πράξεις που επιβάλλονται σε σχέση με την ε, κοινή εργοτική πολιτική και τη μεταρρύθμισή τη. Έχουμε φτάσει σε ένα στάδιο μάλιστα που κάποιοι ευρωβουλευτέ λένε ότι προτιμούν να ασκήσουν βέτο και να μην υπάρξει καθόλου μεταρρύθμιση τη ε, ΚΑΠ παρά να ε, κάνουν πίσω σε σημεία που θεωρούν σημαντικά και πολύ αρνητικά. Υπάρχει λοιπόν ε, σημαντικός αναβρασμός ε, σε ό,τι αφορά το Κοινοβούλιο. Μέχρι τώρα δεν ακούσαμε αντιδράσεις του Συμβουλίου απέναντι στις, στη δική μας συμπεριφορά. Εσείς φαντάζομαι αφού γκράζεστε ως τμήμα της και μέλος της ελληνικής διοίκησης. Ξέρετε ότι και ο υπουργό σα θα προεδρεύσει του Συμβουλίου Γεωργίας. Ποια είναι η δική σας άποψη λοιπόν και η άποψη του Συμβουλίου ε, αγανακτή με τη συμπεριφορά του Κοινοβουλίου. Θα θέλαμε να μάθουμε μερικά πράγματα παραπάνω για τις δικές σας απόψεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντέ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητέ συνάδελφε, κύριε Σταμενίτη, σας ευχαριστώ που ήρθατε. Θέλω να υπογραμμίσω και εγώ αυτά που είπε η συνάδελφος Εράντς ήδη. Ο κύριος Παπαστάνκος μας ενημέρωνε ανέκαθεν ε, για την κατάσταση ελληνικής γεωργίας και πραγματικά θα χαρούμε ε, πάρα πολύ αν βελτιωθεί η υγεία του ε, και σύντομα. Θέλω να ρωτήσω κάτι ως προς την αισιοδοξία σας. Είπατε με αισιοδοξία ότι εφαρμόζεται η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Εγώ ανησυχώ βαθύτατα. Έλαβα μια επιστολή από τη γερμανική διοίκηση πριν από λίγο που αναφέρεται στην υλοποίηση του Ταμείου για τη Θάλασσα και την Αλία και εκφράζουν σφοδρότατες ανησυχίες για τη γραφειοκρατία που θα χρειαστεί στο μέλλον για να εφαρμοστεί αυτό. Στο παρελθόν όταν κάποιος ζητούσε 2.000 ευρώ έπρεπε να απαντήσει περίπου σε 30 ερωτήσεις. Με τη νέα πράξη που έχει καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι 100 οι ερωτήσεις για να πάρεις μια επιδότηση 2.000. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε φορά μιλάει για κατάργηση της γραφειοκρατίας και με κάθε νέο κανονισμό έχουμε περισσότεροι και όχι λιγότεροι. Και αν γίνει το ίδιο με το Ταμείο για τη Θάλασσα και την Αλία και αυτό μεταφερθεί και στη Γεωργία, τότε θα έχουμε ένα γραφειοκρατικό τέρας ε, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης κοινή γεωργικής πολιτικής. Ε, όλα αυτά τα μέτρα, το πρασίνισμα, το ένα, το άλλο, ανησυχώ πάρα πολύ για τις ε, κατεξιοδότηση πράξεις, για τις προθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέχρι τώρα μόνο ε, συντακτικές διορθώσεις και βελτιώσεις στη διατύπωση μας έχει στείλει. Και το λέω ρητά, αν θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόσει ως έχουν τις κατεξοδότηση πράξεις, δεν πρόκειται εγώ ποτέ να τις υπερψηφίσω. Θα ζητήσω και ονομαστική ψηφοφορία και το δικό μου όνομα δεν το βάζω κάτω από τέτοια γραφειοκρατική εφαρμογή με εκπλήσει η αισιοδοξία σας. Πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει στο Συμβούλιο να προσέξουν πάρα πολύ τι τους περιμένει γιατί για την εφαρμογή και την υλοποίηση όλων αυτών θα είναι αρμόδια τα ίδια τα κράτη-μέλη στη συνέχεια. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Καπούλα Σάντος, θα ήθελα να καλωσορίσω τους επισκέπτες του μια ομάδα επισκεπτών και να σας πω ότι ο κύριος Καπούλας ήταν και ε, εισηγητή σε δύο σημαντικές εκθέσεις ε, για την μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Και αν πάει κάτι στραβά, ξέρετε τι σπταίει, ποιο να κυνηγήσετε ε, όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τον φιλοξενούμενό μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ζητώ συγγνώμη που δεν άκουσα όλη την παρέμβασή σας, αλλά όπως είπε και ο Πρόεδρος, ήμουν σε μια συνεδρίαση, είχα συνάντηση με διαφόρους εκπροσώπους συνεταιρισμών της Πορτογαλίας που ήρθαν εδώ σήμερα και παρακολουθούν από κοντά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η κοινή αγροτική πολιτική και πώς εφαρμόζεται στην Πορτογαλία. Ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τη δική σας αξιολόγηση, κύριε Σταμενίτη, για το τελικά αποτελέσματα και τις προοπτικές της εφαρμογής της ΚΑΠ ε, στην Ελλάδα. Συμμερίζομαι πολλά από τα σχόλια που άκουσα να εκφράζετε. Πράγματι είναι ζωτική σημασία για μα να συνεχίσουμε να έχουμε μια κοινή αγροτική πολιτική στην Ευρώπη. Είναι θέμα συνοχή. Μα βοήθησε να καταπολεμήσουμε τη φυγή από την Ήπεθρο. Κρατά τον κόσμο στην Ήπεθρο με οικονομική δραστηριότητα. Έτσι γινόμαστε ανταγωνιστικοί. Και έτσι η Ευρώπη παραμένει με σημαντικός εξαγωγέας, μεγάλος εξαγωγέας αγροτικών προϊόντων. Συμφωνώ με τα σχόλιά σας. Έρχομαι τώρα, ερχόμαστε σε ένα στάδιο μάλλον, πέρα από αυτό που αναφέρθηκε για τις κατεξοσιοδότηση πράξεις, που υπάρχει αντιπαράθεση μεταξύ Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ελπίζω να επικρατήσει κοινή λογική από πλευράς ε, Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να λάβουν υπόψη κάποιες από τις δικές μας θέσεις, και η πλέον πρόσφατη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πράγματι προβλέπει μεγαλύτερη ευελιξία, όχι αρκετή ακόμα, αλλά χαίρομαι που μπορούμε να βλέπουμε μια κάποια ευελιξία. Όμως πέρα από αυτό, Έχω μία ερώτηση από εσά, συνάδελφε, κύριε Βουλευτά. Ποια είναι η κατάσταση τώρα στην Ελλάδα που επικρατεί όσον αφορά τους ενεργούς γεωργούς. Θα είναι πιο ανοιχτή η Ελλάδα, θα είναι πιο επιλεκτική όσον αφορά τους δικαιούχους που ωφελούνται από την κοινή αγροτική πολιτική και για τους μικρούς γεωργούς επιθελοντικής βάσεως ε, θα το εφαρμόσει αυτό η ε, ελληνική κυβέρνηση για την περιφερειοποίηση των άμεσων πληρωμών. Αυτή είναι μια άλλη ερώτηση. Θα επιλέξει η Ελλάδα περιφερειακή λύση ούτως ώστε να εξασφαλίζει μεγαλύτερη δικαιοσύνη ή θα χορηγείται η ενίσχυση σε εθνικό επίπεδο. Και τέλος, έχω μια ερώτηση για το ελληνικό πρόγραμμα αναπτύξεως της υπαίθρου. Το έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συζητείται ακόμα με τους ε, διαφόρους εμπλεκόμενους φορείς. Θα ήθελα να ακούσω ποιο είναι το εύρος των συζητήσεων στην Ελλάδα όσον αφορά ε, την άποψη των παραγωγών των διαφόρων ενδιαφερομένων. Έχουν συμμετάσχει πολλοί στη συζήτηση για την ανάπτυξη αυτού του προγράμματος για την ανάπτυξη πέθρου. Οποιασδήποτε πληροφορίες μπορείτε να μου δώσετε με τα χαράς να τις ακούσω. Σας καλωσορίζω και σας εύχομαι και σε εσά και στη χώρα σας κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ, λέω ο Πρόεδρος. Εάν δεν υπάρχουν άλλες ε, ερωτήσεις, θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια στο προηγούμενο σημείο που συζητούσαμε στην ημερήσια διάταξή μας. Συζητήσαμε τις διαπραγματεύσεις της συμφωνίας TTIP με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Ακούστηκαν διάφορες ανησυχίες στην Επιτροπή όσον αφορά αυτή την συμφωνία. Αυτό είναι το πρώτο ζήτημα. Και δεύτερον, ποια είναι η κατάσταση τώρα, ποια είναι η κατάσταση για εκείνους που ζουν στην Ήπεθρο, που ασχολούνται με τη Γεωργία. Ποια ήταν η συνέπεια της κρίσης για αυτούς τους ανθρώπους, όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης των αγροτών, ποια είναι η συνέπεια, ποια είναι η κατάστασή τους, ποια είναι η κατάσταση στην Ήπεθρο, ποια είναι η θέση των μικρών γεωργών στη χώρα σας. Ξέρω ότι υπάρχει ένα εισοδηματικό πρόβλημα, εισοδηματική κρίση στην Ελλάδα που έχει σοβαρότατο αντίκτυπο κυρίως για τους μικρούς γεωργούς και θα ήθελα να, σχολιά, να αντιδράσετε στις ερωτήσεις μου, στα σχόλιά μου και στις ερωτήσεις των μελών σας παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ και για τις ευχές που δώσατε για τον συνάδελφό σας, τον κύριο είναι έναν άνθρωπο που γνώρισα πάρα πολύ καλά από το 1990 όταν ήταν υπουργό της κυβέρνησης ε, με τον κύριο Παπαστάνκου οι γενέτειρέ μας έχουν μόνο 30 χιλιόμετρα. Είναι από τη Βέρεια, εγώ κατάγομαι από τα Γενιτσά και οι δύο περιοχές είναι ε, έντονα γεωργικέ ε, περιοχές. Ε, στην περιοχή μα παράγονται ροδάκινα συμπύρινα, μεταποιούνται και γίνεται κομπόστα. Όπως επίσης είναι και περιοχές σημαντικές όσον αφορά την παραγωγή του κερασιού αλλά και άλλων καλλιεργιών όπως είναι το βαμβάκι και το, βαμβάκι και, ε, το καλαμπόκι. Απαντώντας από το τέλος του κύριο Πρόεδρο, θα ήθελα να πω ότι οπωσδήποτε η κρίση στην ελληνική, στην Ελλάδα, επηρέασε και τους ε, αγρότες. Ε, ήταν, θα, θα ήταν αδύνατο να μην τους επηρεάσει. Όμως θεωρώ ότι η εφαρμογή της κοινή γεωργικής πολιτικής που άρχισε την προηγούμενη περίοδο και ολοκληρώνεται το 2013, ήταν ένα σημαντικό όπλο για να προστατέψει αρκετά ε, τους αγρότες. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι η εφαρμογή της κοινή γεωργικής πολιτικής και αυτή που μετεξελίσσεται από το 2015 μέχρι το 2020 είναι ένα σημαντικό όπλο ώστε να μετεξελίξουμε την γενική γεωργία και να δώσουμε όθηση ώστε να υπάρχει μια κινητικότητα από τις δύο μεγάλες πόλεις στην περιφέρεια. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες αγρότες ε, τα ανέφερα επιγραμματικά και στην τοποθέτησή μου είναι αυτό που σας είπα ότι είναι, υπάρχουν μικροί κλήροι και η Ελλάδα είναι μια ορεινή χώρα με διαφορετική ε, όσον αφορά το υδάτινο ισοζύγιο μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Όμως αντιμετωπίζουμε και άλλα προβλήματα και αυτό έχει να κάνει με το υψηλό κόστος ενέργειας. Εκεί είχαν μια σημαντική επιβάρηση οι αγρότες καθώς για να αντιμετωπίσουν τα δημοσιονομικά μας προβλήματα αυξήθηκε κατά πολύ το κόστος πετρελαίου και στη συνέχεια για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του 2020 για την ενέργεια του περιβάλλον αυξήθηκε το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, άρα είχαμε μια επιπλέον επιβάρυνση στους αγρότες το ένα αφορά την κρίση, το άλλο αφορά του σχεδιασμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το περιβάλλον. Και το τρίτο μεγάλο πρόβλημα των Ελληνίων αγροτών είναι αυτή η δυσκολία που υπάρχει με τα φυτοφάρμακα και με τα λοιπάσματα όπου δεν υπάρχει ελεύθερη διακίνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι λοιπόν υπάρχουν άλλε τιμέ στην Ελλάδα, άλλε τιμέ στην Βουλγαρία, άλλε τιμέ στην Ιταλία, χώρε οι οποίε είναι ανταγωνιστικέ τη χώρα μα. έχουμε ακριβά, ακριβότερα εφόδια, γιατί υπάρχει αυτός ο περιορισμός της ελεύθερης διακίνησης. Ανέφερα ποιε είναι οι σκέψει μα. Δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα αυτή, αν επιτρέπεται, η έκφραση τη εθνικοποίηση τη κοινή γεωργική πολιτική στη χώρα μας. Έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα ερχόμαστε και συζητάμε πώ θα την εφαρμόσουμε στη χώρα μας. Οι πασεγέ που είναι το τριτοβάθμιο όργανο των αγροτών έχει κάνει πάρα πολλέ συζητήσει, έχει κάνει πάρα ημερίδε σε όλη την Ελλάδα και βρισκόμαστε μέσα στην επόμενη άνοιξη στο να καταλήξουμε πώ θα εφαρμοστεί αυτή η νέα κοινή γεωρική πολιτική στη χώρα μα. Ανέφερα τέσσερα σενάρια, είναι υποσυζήτηση είναι αυτά, τα επαναλαμβάνω. Ένα μπορεί να θεωρηθεί όλη η χώρα ω μία περιφέρεια ή να χωριστεί η χώρα σε 13 περιφέρειες όπως είναι η διοικητική της διάρθρωση ή σε δύο περιφέρειες καλλιεργούμενων εκτάσεων και δεύτερη βοσκοτόπων και το τελευταίο σενάριο αφορά ε, τέσσερις περιφέρειες όπου έχουμε πρώτον τις καλλιεργούμενες παιδινές, τις καλλιεργούμενες ορεινές, τους βοσκότοπους παιδινών και τους βοσκότοπους ορεινών εκτάσεων. Δεν έχουμε καταλήξει ακριβώς πώς θα δοθούν οι ένες ενισχύσεις και είμαστε μια διαδικασία συζητήσεων. Έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση στη χώρα μας και με τους αγρότες και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αλλά και με την κυβέρνηση. Πάντως, ε, νομίζω ότι θα καταφέρουμε όποιο σενάριο και να επιλεγεί να υπάρχει αυτή η εξισορρόπηση της μοναδίας αξίας δικαιώματος μεταξύ των διοικητικών περιφερειών και ανάμεσα τους παραγωγούς. Θα υπάρχουν κάποιοι παραγωγοί που θα πάρουν λιγότερα χρήματα και κάποιοι θα πάρουν περισσότερα χρήματα γιατί υπήρχε μια ανισότητα στην προηγούμενη κατάσταση. Ε, εμείς ε, έχουμε αισιοδοξία για τη μεταρρύθμιση γιατί η κοινή γεωργική πολιτική μας βοήθησε πάρα πολύ ώστε να σταθούν οι Έλληνες αγρότες στα πόδια τους. Αυτό αισιοδοξούμε ότι θα το κάνει και η νέα κοινή γεωργική πολιτική που ουσιαστικά είναι με συνέχεια της προηγούμενης. Πράγματι υπάρχει γραφειοκρατία η οποία θα αντιμετωπιστεί, αλλά είμαστε εδώ στην χώρα μας να το αντιμετωπίσουμε συζητώντας με την κυβέρνηση πώς ακριβώς θα εφαρμόσουμε αυτά. Ε, πράγματι συζητάμε ακόμα για τους ενεργούς αγρότες, ποιοι είναι, και ποιοι θα είναι οι περιορισμοί. Υπάρχει κυρίαρχη άποψη ότι πρέπει να είναι κατ' επάγγελμα αγρότε αυτοί που θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή την ενίσχυση για να μπορούμε να ενισχύσουμε αυτή την προοπτική και την πολιτική ε, ανάπτυξη υπαίθρου. Εμείς πιστεύουμε ότι στη χώρα μας, πέρα από τον τουρισμό που αποτελεί την αυαρχίδα ε, της παραγωγής στη χώρα μας, ο πρωτογενή τομέα, η γεωργία και η κτηνοτροφία μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο ώστε να μπορούμε να καλύψουμε το εμπορικό ισοζύγιο. Διαθέτουμε σημαντικά προϊόντα όπω είναι το λάδι, οι ελιέ καλαμών, η φέτα, το γιαούρτι, η μαστίχα χαχή, ο κρόκος κοζάνης, αναρρύθμιτα προϊόντα ονομασία προέλευση, τα οποία θέλουμε και να βελτιώσουμε τις ποσότητες και την ποιότητα, αλλά να βελτιώσουμε και τη μεταποίηση αυτών και να βρούμε ενέργειες και δράσεις να προωθήσουμε αυτά τα προϊόντα στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Πιστεύουμε ότι η κοινή γεωρική πολιτική έχει αυτές τις δράσεις, έχει αυτές τις ενέργειες για να μπορέσει να μας βοηθήσει όλους τους γεωργούς, όχι μόνο της Ελλάδος αλλά όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρήσουμε. Γιατί όπως σας είπα και πριν, το μείζον είναι να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα όλοι μαζί. Μόνο ενωμένοι μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με κοινέ πολιτικέ τι οποίε θα συζητήσουμε, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσει που έχουμε σήμερα. ότι... Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο η κατεξοδότηση πράξη και πώ θα αντιμετωπίζει το Κοινοβούλιο είναι κάτι το οποίο μα δίνει. Ε, ε, θεωρούμε καταρχήν ότι είναι θετικό αρκεί να μην, φεύγει, να μην ξεφεύγει από, από την προοπτική της κοινή γεωργικής πολιτικής. Γιατί θα δώσει τη δυνατότητα στη χώρα μας, όπως και σε κάθε χώρα, να εφαρμόσει την κοινή γεωργική πολιτική ε, έχοντας ε, λάβει υπόψη της τις ιδιαιτερότητες και, τις, τη διαφοροποίηση που έχει η γεωργία και η κοινοτροφία σε κάθε χώρα αλλά και σε κάθε διαφορετικό διαμέρισμα της χώρας μας. Αυτό θα δώσει την ευελιξία ώστε να προχωρήσουμε σε αυτό, αρκεί πάντοτε να μην φύγουμε από το κεντρικό στόχο. Και νομίζω εδώ είμαστε και οι Έλληνες βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αλλά και εσείς και οι υπόλοιποι βουλευτές των άλλων κοινοβουλίων, ώστε να ελέγξουμε αυτή την προοπτική. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και τη δυνατότητα που ε, είχα να εκφράσω τις απόψεις και τις σκέψεις και ελπίζω να βοήθησα ελάχιστα έτσι, περισσότερο στο να γνωρίσετε τις σκέψεις μας και πώς είναι οι Έλληνες αγρότες στη χώρα μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ε, παρουσίασή σας ε, και τις απαντήσεις που δώσατε. Είναι μια νέα παράδοση. Συναντούμε ε, μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων της χώρας που ασκεί την Προεδρία. Αυτό βεβαίως μας ωφελεί ιδιαίτερως γιατί έτσι έχουμε μια καλύτερη εικόνα της γεωργίας Τη χώρα ε, που έχει την Προεδρία στα χέρια τη. Και επίσης μα ενδιαφέρει ιδιαίτερω να γνωρίζουμε τι συμβαίνει στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο. Πολύ συχνά πρέπει να σας πω ότι ως μέλη κοινοβουλίων έχουμε περισσότερα κοινά από ότι τα μέλη του Κοινοβουλίου με την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Και πάλι σας ευχαριστώ λοιπόν. Εάν δεν υπάρχει κάποιο άλλο ερώτημα, θα ήθελα να προτείνω ένα σύντομο διάλειμμα του ενός λεπτού για να αποχαιρετήσουμε όλους ε, τους ε, καλεσμένους μας και μετά θα περάσουμε στο τελευταίο σημείο της μέσης διάταξης σήμερα. Ευχαριστώ και πάλι τον κύριο Σταμενίτη και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο σε εσάς και στους συναδέλφους σας. Καλή τύχη λοιπόν, καλή επιτυχία ε, με τις ενέργειές σας προς όφελος της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως η δική μας θητεία λίγη, αλλά έτσι πάνε τα πράγματα στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε πολύ. proszę państwa przechodzimy do ostatniego punktu Συνάδελφοι, τώρα θα περάσουμε στο τελευταίο σημείο της σημερινής τη διάταξης ε, για, τα, για τις ενέργειες ενημέρωση σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα και προώθησής τους θα έχουμε μια νέα, νέα ενημέρωση για την πολιτική προώθηση των ευρωπαϊκών προϊόντων. Πριν δώσουμε λοιπόν το λόγο στην κυρία Χεράς Γκαρσία, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε ένα πολύ αυστηρό χρονοδιάγραμμα εάν θέλουμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη ανάγνωση πριν από τις εκλογές. θα πρέπει να επιδείξουμε επιθαρχία σε ό,τι αφορά την τήρηση του αυστηρού αυτού χρονοδιαγράμματο. Λοιπόν, η προθεσμία υποβολή ε, τροπολογιών 14 Φεβρουαρίου στι 12 το μεσημέρι. Μέχρι τότε έχετε περιθώριο να υποβάλλετε τροπολογίε. Η κυρία Χεράν Γκαρσία έχει τον λόγο. Πολύ ωραία το είπατε, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Και Μ' αρέσει που μου λέτε το όνομά μου σωστά, γιατί και η κυρία Γκαρσία από του σοσιαλιστέ είναι σκιώδη συγγήτρια. Λοιπόν, τώρα σοβαρά. Πραγματικά αυτό το έγγραφο είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, και το ζητάει ο κλάδος, η ε, ε, γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι και οι εργαζόμενοι στην τροφιμική βιομηχανία. Χρειαζόταν λοιπόν να έρθει αυτό το έγγραφο για προώθηση των τροφίμων μας. Μας έχουν διαβιβάσει λοιπόν την ανάγκη αυτή και την επιθυμία οι αγρότες εδώ και καιρό. Επιθυμούν διακαώς να κάνουμε ό,τι μπορούμε και γρήγορα ε, για να εγκριθεί αυτό το κείμενο. Θα μπορούσε να είχε έρθει πολύ νωρίτερα, εν πάση περιπτώσει τώρα το λάβαμε και πραγματικά ενδιαφέρονται πολύ περισσότεροι να εγκριθεί σε πρώτη ανάγνωση το συντομότερο το θέλει ο κλάδος και ο Επίτροπος ενδιαφέρεται πάρα πολύ να εγκριθεί σε πρώτη ανάγνωση και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε εμείς ό,τι περνάει από το χέρι μας για να γίνει αυτό και να είναι όσο γίνεται πιο συντονισμένη η συνεργασία μας με τις πολιτικές ομάδες. Ωραία, έρχομαι τώρα στην ουσία του κειμένου. Σήμερα οι πολίτες ε, αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερο σκληρό ανταγωνισμό και ανελαίητο από τις τρίτες χώρες. Και ξέρουμε ότι οι διακοιμάνσεις των τιμών είναι πολύ μεγάλες, το γνωρίζουμε. Γι' αυτό χρειάζεται βελτίωση ο ισχύων κανονισμός για τις εκστρατείες ενημέρωσης και προώθησης των γεωργικών μας προϊόντων. Αυτό τον καιρό γίνονται διαπραγματεύσεις, όπως μας είπε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με σημαντικές τρίτες χώρες. Είπα, Μερκοσούρ και θα πρέπει να αναδείξουμε και πάλι την παραγωγή μας για να μπορούν τα προϊόντα μας να ανταγωνίζονται. Είναι πολύ χρήσιμες αυτές οι εκστρατείες και οι καμπάνιες για την κρίση ε, που προκύπτει μετά από μείωση των τιμών ή επιζωοτίες ή άλλα προβλήματα υγείας. Θυμάστε το σκάνδαλο με την εσερίχια κόλλη, το κολοβακτηρίδιο όπου είδαμε η πρόθεση πώς μπορεί να χρησιμοποιείται με τρόπο πολύ ευέλικτο, πολύ περισσότερο από ό,τι σήμερα. Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πολύ περιορισμένη δυνατότητα πρωτοβουλίας, όπως φάνηκε άλλωστε, όταν ξέσπασε αυτή η κρίση για να μην αντιμετωπίζει τέτοιου είδους κρίσεις και δεν έχει καμία την παραμικρή πρωτοβουλία για να ξεκινήσει προώθηση και ενημέρωση σε περίπτωση κρίσης στην αγορά που δεν έχουν οι κρίσεις αυτές υγειονομική προέλευση. Το άρθρο 45 του χρηματοδοτικού προϋπολογισμού, ε, κανονισμού συγγνώμη, της ΚΑΠ προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενημερώνει όταν χάνει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε κάποια προϊόντα. Όπως είδαμε και στην περίπτωση του κολοβακτηριδίου ε, σε ρίχια κόλλη, είναι πολύ περιορισμένες σε εμβέλεια αυτές οι δράσεις και πολύ μικρός ο προϋπολογισμός. Και ε, τότε ελήφθησαν κάποιες ε, δράσεις, ε, μετά από πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά πέρασαν σχεδόν απαρατήρητες. Σήμερα δεν υπάρχει καμία νομική δυνατότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ενημέρωση και προώθηση μετά από διάφορες κρίσεις, διαφορετικές επαναλαμβάνω από υγειονομικές, ας πούμε κρίση αγοράς που είδαμε στα γαλακτοκομικά ε, πριν από λίγο καιρό. Δεν υπήρχε κάλυψη για αυτή. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια επίκουσα διαδικασία για την ενημέρωση και την προώθηση όταν έχουμε κρίσεις υγειονομικές ή ε, αναταράξεις στην αγορά και να μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα ε, λαμβάνει αυτά τα μέτρα ιδία πρωτοβουλία. Ελπίζω να μην διαφωνήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμεί θέλουμε να του δώσουμε περισσότερη εξουσία απέναντι σε κρίσιμε καταστάσει. Εδώ και καιρό η κοινή γεωργική πολιτική, όπω σα είπα και προηγουμένω, στερείται αυτή τη δυνατότητα προώθησης ε, των γεωργικών προϊόντων. Γι' αυτό ε, γνώρισε τέτοια υποδοχή. Προβλέπει και αύξηση του προϋπολογισμού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από 61,5 εκατομμύρια στα 200 εκατομμύρια το 2020. Καταλαβαίνετε εδώ ποια είναι η πρόθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ποντάρει σοβαρά σε αυτό το εγχείρημα. Ποιο είναι, ποια είναι η μεγάλη καινοτομία τα εμπορικά σήματα και η προέλευση των προϊόντων. Αυτά τα δύο εντός των δράσεων που θα χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν από τις βασικές ε, διεκδικήσεις του κλάδου, διότι αν δεν υπήρχαν αυτά τα δύο στοιχεία δεν θα μπορούσαμε ε, να έχουμε τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της χρηματοδότησης για τους κλάδους που θίγονται. Θα πρέπει να ενισχυθεί, να αναβαθμιστεί ε, το προϊόν, αυτό δεν είναι μόνο υπέρ της συγκεκριμένης μάρκας του εμπορικού σήματος, αλλά θα συμπαρασύρει και άλλες μάρκες ε, μαζί της ε, όταν προωθηθεί αυτή. Όταν υπάρχει αρκετή κάλυψη, ξέρω ότι ορισμένοι το βλέπετε επικριτικά, αλλά σας λέω να σκεφτείτε, μια γνωστή μάρκα, ένα ε, μεγάλο εμπορικό σήμα συμπαρασύρει και βοηθάει και λειτουργεί ως ομπρέλα και για άλλα προϊόντα, για άλλες μάρκες λιγότερο γνωστές θα ήταν λίγο ωφελές από πλευράς μου να θεωρήσω ότι οι περιορισμοί ε, που επιβάλλονται ε, θα έφταναν από μόνοι τους για να αντιμετωπίσουν ε, την έλλειψη και την απώλεια εισοδήματο. Δεν είναι καμία πανάκια, ούτε το ισχυρίζομαι, αλλά θα βοηθήσουν και απέναντι σε διαπραγματεύσεις, όχι μόνο με τις ΗΠΑ Πολιτείες που ακούσαμε σήμερα, αλλά και τις υπόλοιπες η πρόθεση των ευρωπαϊκών προϊόντων είναι πάρα πολύ σημαντική και σε αυτό το κλάδο επίσης στο πεδίο θα πρέπει να είναι ενήμερος ο Ευρωπαίος καταναλωτής για τα ίδια χαρακτηριστικά της παραγωγής μας αλλά και για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων θα πρέπει να γνωρίζουμε τι προσπάθειες καταβάλουν οι Ευρωπαίοι ε, παραγωγοί για τα προϊόντα, για την προστασία του περιβάλλοντος, για τη βελτίωση της υγείας και αυτά να γίνονται γνωστά και εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, να υπάρχει πιο απλή διαχείριση απέναντι σε τρίτες χώρες και αυτή μεγάλη καινοτομία και πρόοδος την κεντρική διαχείριση θα έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω αυτό θα λύσει κάποια προβλήματα συντονισμού που ανεκύψαν στο παρελθόν μεταξύ των κρατών μελών. Για τα ποσοστά, πόσο θα πρέπει να αφιερώνεται για το εξωτερικό και πόσο για το εξωτερικό της Ένωσης. Θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι η βασική αγορά μας είναι η εγχώρια. Αλλά επίσης θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι έχουμε και μεγαλύτερο δυναμικό προς τα έξω. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε πού χρειάζεται περισσότερη στήριξη των παραγωγών απέναντι στην εξωτερική απειλή ας πούμε ή τον εξωτερικό ανταγωνισμό αλλά να δούμε και στο εξωτερικό πώς μπορούμε να προωθήσουμε τα προϊόντα μας. Δεν ξέρω, 75, 25, 60, 40 θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό. Η εθνική συγχρηματοδότηση αποκλείεται ε, από τα μέτρα αυτά αυτό ανησύχησε πάρα πολύ τους ενδιαφερομένους και μεταξύ αυτών και συναδέλφους. Ε, γιατί, διότι ο κλάδος ανησυχεί ότι θα συμμετέχει περισσότερο ο ίδιος οικονομικά, ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι εταιρείε αυτές ε, που παράγουν τρόφιμα έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση όπως όλες οι επιχειρήσεις για να μην πω και περισσότερο. Όταν εκπονήθηκε η έκθεση αυτή, κατά τη διάρκεια της εκπόνησης ε, λάβαμε πολλές αντιρρήσεις για την κατάργηση αυτή της εθνικής χρηματοδότησης που είναι θελούσια. Εγώ κάνω γενικά τροπολογίες για την αύξηση της χρηματοδότησης και της κρατικής και να μπουν ε, συγκεκριμένες διατάξεις και προβλέψεις για τομείς πάρα πολύ ευαίσθητους ε, όπως είναι ο γαλακτοκομικός. Η πρόταση ευρωπαϊκή Επιτροπής δίνει τη δυνατότητα να χρηματοδοτούνται τα ε, προϊόντα του πρώτου παραρτήματος και ορισμένα άλλα μεταποιημένα τρόφιμα. Εγώ πάω ακόμα παραπέρα. Γιατί να περιοριστεί ο κατάλογο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν το δικαιολογεί. Γιατί το προτείνει αυτό το κατάλογο ε, που είναι περιοριστικό. Κατά το δοκούν, μ' αρέσει αυτό το προϊόν, το άλλο δεν μ' αρέσει. Όχι. Θα πρέπει να αφήσουμε αυτό ανοιχτό και σε άλλα προϊόντα. Χωρί να εξαιρείται κανένα τομέα. Βέβαια, να έχουμε κάποιε περιοριστικέ διατάξει που να ε, ενισχύεται περισσότερο και κατά προτεραιότητα ο πρωτογενής τομέας. Γνωρίζουμε μια μεγάλη οικονομική κρίση αυτό τον καιρό και δεν θα πρέπει να ε, κάνουμε παζάρια τώρα ε, τσιγκουνιές. υπάρχουν πολλά προϊόντα που τα γνωρίζει ο καταναλωτή και να ενισχύονται και να προωθούνται και οι μάρκες, είπαμε, οι οποίε θα συμπαρασύρουν και άλλα εμπορικά σήματα. Θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριληφθεί και ο ίνος εδώ και να βελτιωθεί η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο ίνος είναι από τα προϊόντα, ακριβώ αυτά που σα λέω, ομπρέλα, που από κάτω θα μπορούσαν να ενταχθούν πολλά άλλα προϊόντα. Είναι ένα προϊόν πάρα πολύ γνωστό, είναι ένας από τους τομείς που μας ενδιαφέρει ε, περισσότερο και μας εκπροσωπεί σκοπεύει εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δίνει μια εικόνα για τα τρόφιμα και τον πολιτισμό μας και θα πρέπει να είναι στην ίδια μοίρα και επίσης όρις να αντιμετωπίζεται. Δεν θα πρέπει να εξαιρείται λοιπόν το κρασί από τη δυνατότητα συμμετοχής σε αυτές τις εκστρατείες. Μόνο του ή και με άλλα. Εκτελεστικοί οργανισμοί. Γιατί να μην το αναλαμβάνουν. Αν υπάρχει ένα τέτοιο όργανο που μπορεί να το αναλάβει, γιατί όχι. Εμείς δεν θέλουμε να αυξηθεί η γραφειοκρατία, η διοίκηση, αλλά με τα δεδομένα μέσα και πόρους να προχωρήσουμε. Αυτός ο οργανισμός θα μπορούσε να παρέχει και τεχνική υποστήριξη και αρρωγή στους ε, φορείς, δηλαδή παροχή συμβουλών και βοήθεια για να βελτιώνονται η προστασία των ευρωπαϊκών προϊόντων απέναντι σε ε, απομιμήσεις και παραποιήσεις, μαϊμού δηλαδή προϊόντα από τρίτες χώρες. Επίσης δεν θα πρέπει οι εθνικές διοικήσεις να είναι άμυρες ευθυνών, γιατί αυτές τελικά το αναλαμβάνουν, θα πρέπει να έχουν λόγο. Και ε, επίσης θεωρώ πάρα πολύ καλή την πρόταση ενός προγράμματος εργασίας, γιατί αυτό θα μας δίνει σαφείς στρατηγικέ. Ποιος είναι ο στόχος, τι θέλουμε να πετύχουμε και επί μια τριετία, τριετία, διότι θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι τριετές το κάθε πρόγραμμα τόσο διαρκούν οι εκστρατείε εκστρατείες προώθησης. Τριετία. Ε, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χωράει βελτίωση και το κάνω και στο κείμενό μου. Θα πρέπει να συμπεριλάβουμε ένα κατάλογο σαφών και συγκεκριμένων στόχων που καλείται να καλύψει αυτό το πρόγραμμα. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να περιορίσει τη δράση της σε αυτό που ε, αναφέρεται στη βασική πράξη. Τώρα, στη διάκριση που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χώρη αγορά και αγορά τρίτων χωρών, νομίζω ότι αυτό θα κάνει τα πράγματα πιο άκαμπτα. Προσπάθησα να τα ενώσω και τα δύο, διότι θα πρέπει να είναι ενιαία η ταξινόμηση των δράσεων που μπορεί κανείς να χρηματοδοτεί εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Οι ε, εκστρατείες προώθησης έτσι δεν αποκλείονται από την εσωτερική αγορά, όπως σας είπα προηγουμένως, και θα πρέπει να ενημερώνται οι καταναλωτές και τρίτων χωρών για τις υψηλές ε, προδιαγραφές ποιότητας που καλύπτει η κοινοτική παραγωγή. Ενισχύουμε λοιπόν τα όσα ήδη κάνουν οι παραγωγοί μας. Αυτά σε γενικές γραμμές είναι η πρόταση του, κανονισμού, του της έκθεσης συγγνώμη, ε, περιμένω τα σχόλιά σας και θέλω να τελειώσω την παρέμβαση λέγοντας ότι πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος. 14 του Φλεβάρι πρέπει να έχουμε τις τροπολογίες, θα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ γρήγορα και ελπίζω να συνεννοηθούμε πολύ γρήγορα και να τα βρούμε με τους κοιόδης ηγητές και τους υπολείπους συναδέλφους που ενδιαφέρονται. Όποιος θέλει μπορεί να συνεργαστεί σε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Αγιούσο και μετά η κυρία Μαγκίνας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μήπως πρώτα να μιλήσεις και όδηση ηγήτρια της άλλης πολιτικής ομάδας. Εγώ με χαρά να μιλήσω, αλλά θέλω να ακούσω πρώτα την κυρία Γκαρσία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Αγιούσο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για να είμαι ειλικρινής, αυτά που λέγει η συγγήτρια για την ανάγκη επιτάχυσης όσο γίνεται των χρόνων για να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό αυτή η προσπάθεια είναι κάτι που συμμερίζομαι και εγώ προσωπικά και η πολιτική μου ομάδα. Θέλουμε γρήγορα να προχωρήσουμε. Είναι γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της θητείας αυτής έχουμε κάπως απορροφηθεί από τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωρικής πολιτικής που αφοσιωθήκαμε, αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα πολύ σημαντικά. Αυτό το θέμα της πρόθεσης των ευρωπαϊκών προϊόντων είναι εκ των όνων ουκάνευ και αναδεικνύει ακριβώς την περίφημη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία με τις ε, ποιοτικέ προδιαγραφές που έχουμε, τις τόσο υψηλές και θα πρέπει αυτό να διαβιβάζεται και να μεταφέρεται και στον κόσμο με τη συγκεκριμένη προώθηση. Και γι' αυτό ελπίζουμε το συντομότερο να προχωρήσει αυτή η δουλειά ε, και να χρησιμοποιήσουμε το μέσον αυτό. Σε προηγούμενες ε, συζητήσεις ε, είδαμε να διασκεδάζονται και να διαλύονται ορισμένε ανησυχίε και επιφυλάξει που είχαμε. Ο προπολογισμό, το είπε η κυρία Εράντ, η αύξησή του. Γιατί είχαμε κάποιε αμφιβολίες αν θα ήταν επαρκή ή αυτός ο οργανισμός που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρηματοδοτείται από εκεί. Επενεύει ο Επίτροπος, ε, παρενεύει εδώ στην Επιτροπή μας και μας είπε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ωραία. Τελικά θα έχουμε όλους αυτούς τους πόρους στη διάθεσή μας και ε, χρειαζόταν αυτή η διευκρίνηση. Ως προς το περιεχόμενο των ε, τροπολογιών που ανέφερε η συγγήτρια, συμφωνώ περίπου 100% με τα θέματα που είπε. Υπάρχουν ορισμένα που είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα πρέπει να μπουν οπωσδήποτε όπως αυτό το θέμα της ε, συμπερίληψης του ίνου είναι απολύτως απαραίτητο ή άλλο να διευρυνθεί η συγχρηματοδότηση για ε, προγράμματα που αφορούν περισσότερες χώρες. Ε, έχει καλυφθεί λοιπόν αυτό και κάθε ανησυχία ή επιφύλαξη που θα μπορούσα να έχω εγώ ε, οπότε δεν θα επιμείνω παραπάνω, απλώς επευκαιρία να πω ότι θέλω να ακούσω την ε, άποψη Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μια που παρευρίσκεται, να μας πει τη φρονή για το κείμενο της κυρίας Εράντς. Δεν αμφιβάλλω ότι εάν συμφωνήσει η Επιτροπή μας μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι επόμενες εργασίες διαπραγμάτευσης θα είναι πάρα πολύ ευκολότερες για να μπορέσουμε το συντομότερο να φέρουμε σε αίσιο πέρα σε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζητώ συγγνώμη που έκανα λάθος. Η κυρία Γιούζα έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια καθώς και τη σκιώδη εισηγήτρια γιατί η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν καλή αλλά βελτιώθηκε πρέπει να πω πολύ ουσιαστικά από την έκθεση που κατατέθηκε. Είναι άψογη η έκθεση, καλύπτει όλα τα κενά που ενδεχομένως να υπήρχαν ε, στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο μέλλον δεν θα πρέπει να κάνουμε πολλές τροπολογίες, δεν χρειάζεται. Έχουν καλυφθεί όλοι οι φόβοι, ανησυχίε και προβλήματα που ενδεχομένως να είχαν ανακύψει και δεν είχε λάβει υπόψη της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλω μόνο να επιμείνω και να επενέσω όλος ιδιαιτέρως τις τροπολογίες που έγιναν στο άρθρο 5 στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διεύρυνση του καταλόγου προϊόντων, των επιλέξιμων προϊόντων, συμφωνούμε απολύτως, καθιστά πιο ευέλικτη την έκθεση και ανοίγει και πολλές πόρτες αυτό. Επίσης θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας το εξή. Αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι μόνο η ευρωπαϊκή προσφορά στο σύνολό της, αλλά πρέπει να προσφέρουμε και άλλα προϊόντα που δεν είναι ευρωπαϊκά αλλά που αποκτούν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Όπως είναι ο Ιταλικός καφές, η η Βελγική σοκολάτα ε, και μπορούν να προωθηθούν σε τρίτες χώρες χωρίς να είναι αμυγός και πρωτογενός και αυστηρά ευρωπαϊκά προϊόντα, αλλά απέκτησαν την προστιθέμενη αξία τους από την επεξεργασία στην Ευρώπη. Έτσι προβάλλουμε τα προϊόντα μας και κάνουμε μάρκα, σήμα εμπορικό την ευρωπαϊκή ποιότητα. Πρέπει να σας πω ότι όλες οι τροπολογίες με βρίσκουν σύμφωνοι. Είναι πάρα πολύ ωραία η έκθεση στο σύνολό της. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Μακίνες έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για τη δουλειά που έκανε. Συμφωνώ με τις τροπολογίες σας για την εθνική συγχρηματοδότηση. Είναι πραγματικά σημαντικό αυτό. Σε υποστηρίζουμε εκεί και πολύ και ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να εμπλέκονται κάπως ούτως ώστε όταν χειρίζονται το πρόγραμμα να είχαν κάποια συμβολή στην διαμόρφωσή του πριν το εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει και ευρύτερο θέμα. Όταν σκεφτόμαστε την ποιότητα, καμιά φορά έχουμε υπόψη μας μόνο προϊόντα με ονομασία προέλευσης. Και αυτό είναι ένα μικρό ποσοστό της ε, αγοράς μας των τροφίμων. Δεν είμαι σίγουρη αν καλύπτουμε πλήρως το θέμα των σχημάτων, των προγραμμάτων εξασφάλισης ποιότητας στα κράτη-μέλη. Στην Ιρλανδία θα εστιαζόμασταν στο βόλιο που παράγεται βιώσιμα με χαμηλό ίχνος ε, διοξιδίου του άνθρακος και δεν πρέπει να αποκλείσουμε αυτά τα προϊόντα να μπορούν να καλύπτονται από το όλο πρόγραμμα. Θα ελέγξω τις λεπτομέρειες για να είμαι σίγουρη ότι πράγματι μπορεί να γίνει αυτό διότι στο κάτω-κάτω εγκρίναμε μια μεταρρύθμιση της κοινή αγροτικής πολιτικής με κάπως μειωμένο προϋπολογισμό και μεγαλύτερες απαιτήσει από τους ε, γεωργούς. Έχουμε και εμπορικές συμφωνίες διμερείς που αναμένονται, που θα έχουν αντίκτυπο σε επίπεδο εκμεταλλεύσεων και πρέπει να δώσουμε στους παραγωγούς τη δυνατότητα να πολλούν εκτός και εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και μετά την κατάρριξη των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Είναι επίκαιρη έκθεση και σας εύχομαι να περάσει το σύστημα το ταχύτερο δυνατόν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Μόνο μία τροπολογία θα έχω κατά λοιπά. Είμαι πολύ ικανοποιημένη από την έκθεση αυτά και ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και ο Σκάπουλα Σάντος. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτριά μας, λέει ο κ. Σκάπουλα Σάντος. Έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά και όσον αφορά την ενημέρωση και την προώθηση των, προϊόντων των γεωργικών εντός και εκτός ε, Ευρωπαϊκής Ενώσεως ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο την εποχή της κρίσης και η Γεωργία μπορεί να μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε την κρίση. Υποστηρίζω λοιπόν αυτά που είπε η σκιώδηση συγκήτρια, δηλαδή πρόκειται περί καλής ε, εκθέσεως σίγουρα Κάποιες τροπολογίες ίσως βοηθήσουν, ίσως βελτιώσουν το κείμενο περαιτέρω, όμως αυτό που είπε η συγγήτρια περί αφαιρέσεως των ποσοστών για την πρόθεση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά είναι κάτι που εγκρίνω. Νομίζω ότι προχωράει πολύ μακριά από τις Ευρωπαϊκές Επιτροπές. Θέλουμε να πουλάμε σε τρίτες χώρες, αλλά η εσωτερική αγορά είναι σημαντικότατη για κάποια προϊόντα και υπάρχει τεράστιο δυναμικό που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Εν γέννη λοιπόν υποστηρίζω τις προτάσεις σας κυρία Συγήτρια και ελπίζω ότι είναι αρκετά ισχυρή θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ούτω ώστε να οδηγηθεί σε αποδοχή από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, η έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νίκολσον έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για αυτή την έκθεση. Βεβαίω και υποστηρίζω τον στόχο τη μεγιστοποίηση τη εξαγωγή γεωργικών προϊόντων, ιδιαίτερω προ τι αναπτυσσόμενε τρίτε χώρε και αγορέ εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ νομίζω ότι η Ευρώπη μπορεί να έχει προσταθέμενη αξία και μάλιστα να μεγιστοποιήσει αυτό το όφελος Ίσως όμως αυτή η έκθεση να μας απομακρύνει από αυτό το στόχο. Έχω κάποιε σοβαρές επιφυλάξεις εδώ. Όπως ανέφερα, η, έκθεση της, η πρόταση της Επιτροπής είναι ε, πολύ καλή κατά τη γνώμη μου. Βεβαίως υπάρχουν κάποια σημεία όπου οι, κάποιες τροπολογίες θα μπορούσαν να βελτιώσουν την πρόταση. Στηρίζω πλήρως ε, την πρόταση για το 75% της χρηματοδότησης για τις εξωτερικές ε, αγορές με προπολογισμό μέχρι τα 200 εκατομμύρια μπορούμε να διατηρήσουμε τα τρέχοντα επίπεδα ε, ενημέρωσης και να αυξήσουμε τις δαπάνες κατά 75%. Είναι πολύ σημαντικό τα εθνικά καθεστώτα ποιότητας να μην τίθενται ένα ε, αμφιβόλο από αυτές τις διατάξεις. Σε εθνικό επίπεδο έχουμε πολύ επιτυχημένες εκστρατείες που αυξάνουν ακριβώς αυτή την προσταθμένη αξία που θέλουμε να επιτύχουμε ε, στα κράτη-μέλη και αυτό μπορεί να συνεχιστεί. Στηρίζω την πρόταση της συγγήτριας να έχουμε ξεκάθαρους ε, στόχους για την Επιτροπή. Ποιο πρόγραμμα ε, θέλουμε να έχουμε στο πλαίσιο της βασικής πράξης. Ξέρετε ότι στην βιομηχανία των γεωργικών τροφίμων και της εξελίξεις που υπάρχουν σε αυτόν τον κλάδο μετά από την οικονομική κρίση, ιδίω στη χώρα μου, ήταν ένας από τους κλάδους που επλήγει σε μεγαλύτερο βαθμό. Που ήταν ένας κλάδος που δημιουργούσε ε, που πάντα παρήγαγε πλούτο και θέσει εργασία. Επομένω, ε, σίγουρα θεωρώ ότι πρέπει να συμπεριλάβουμε τα μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα στον κανονισμό. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε τη θέση ε, για τα φορολογικά μέσα για κάποιες ε, οργανώσει, γιατί μπορεί αυτό να επηρεάσει τι χρηματοδότητε με τα κράτη-μέλη. Και όλα αυτά θα πρέπει να τα εξετάσουμε στο πλαίσιο αυτή τη πρόταση. Να είμαι ειλικρινή εδώ, να σα πω με απασχολεί το γεγονό ότι ε, κινδυνεύουμε να το να να πάμε πολύ βιαστικά στην Ολομέλεια και υπάρχει ο κίνδυνος να μην ε, επιδείξουμε την απαραίτητη επιμέλεια σε ό,τι αφορά αυτή την πρόταση. Ως εισηγητής γνωρίζω πόσο καιρό παίρνει η μετάφραση των τροπολογιών και το καθεξής είμαι διατεθειμένος να σας βοηθήσω με κάθε δυνατόν τρόπο, όμως πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι δεν θέλω να κινηθούμε βεβαιασμένα εάν αυτό δεν είναι απαραίτητο, μόνο και μόνο για να μπει ε, μέσα στο καταστατικό μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, πράγματι θα επανέλθω σε αυτό το σημείο. Ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Ρουμπρίξη. Ευχαριστώ. Κατά μία έννοια συμφωνώ με αυτή την ε, έκθεση και στην ομάδα μου το έχουμε συζητήσει και θα τη στηρίξουμε. Ωστόσο, πρέπει να πω ποιος είναι ακριβώς ο απότερος στόχος αυτής της έκθεσης. Τι θέλουμε να επιτύχουμε. Θέλουμε να διαφημίσουμε τα προϊόντα μας ούτως ώστε να ε, στην εσωτερική αγορά ή σε τρίτες χώρες. Η διαφήμιση δεν φτάνει για να το κάνουμε αυτό. Για παράδειγμα, στη χώρα μου, στη Λετωνία, έχουμε έναν αρκετά ανεπτυγμένο κλάδο βιολογικής καλλιέργειας. Βιολογικό ψωμί, διάφορα τυριά και το καθεξής. Όμως όταν πάει κάποιος ε, στα καταστήματα θα δει ότι δεν τα αγοράζουν πολλοί καταναλωτές. Όχι επειδή εμφιβάλλουν για την πολύ καλή ποιότητα των βιολογικών ε, προϊόντων, απλά και μόνο επειδή δεν ε, έχουν τα χρήματα για να τα αγοράσουν. Η κρίση είχε αντίκτυπο και σε αυτό το τομέα. Η Λετωνία μπήκε στην Ευρωζώνη και όλα τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι τιμές ε, των καταναλωτικών προϊόντων έχουν αυξηθεί δραματικά, ενώ δεν έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο με τους μισθούς. Μπορεί κάποιο να πει ότι είναι διαφορετικό το θέμα, όμω καλό θα ήταν το Κοινοβούλιο να εξετάσει και αυτό το ζήτημα. Ε, δεν φτάνει μόνο να διαφημίσουμε τα προϊόντα στην εσωτερική αγορά. Δείτε για παράδειγμα την Κίνα. Έχουν ένα κρατικό πρόγραμμα για την αύξηση της ε, οικονομικής ευημερίας ε, στο σύνολο της επικράτειάς τους. Όμως εδώ στην Ευρώπη Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Θυμάμαι πριν από μερικά χρόνια είχαμε όλα αυτά τα πολύ καλά σχέδια για τις ε, τιμές ε, που εξασφάλιζαν οι γεωργοί. Όμως δυστυχώς ε, οι μεγάλοι παίχτες στην αγορά όπως τα σούπερ μάρκετ είναι αυτοί που καθορίζουν και επιβάλλουν τις τιμές. Και έτσι έχουμε το λεγόμενο dumping των τιμών. Γνωρίζουμε για παράδειγμα, το προϊόν για να φτάσει από την μονάδα καλλιέργειας μέχρι στον ε, χώρο τελικής μεταπόλησης ε, περνάει από πολλά στάδια. Και έτσι πολλοί γεωργοί εξαιτία όλων αυτών των διαμεσολαβητών δεν καταφέρνουν να βγάλουν τα προς το ζήν. Θα τα εξετάσουμε πολύ λεπτομερώς όλα αυτά τα σημεία στο μέλλον. Η κοινή γεωργική πολιτική. Μας έδωσε την χρηματοδότηση, χαμηλή χρηματοδότηση βεβαίως για την επόμενη θητεία, όμως εδώ βλέπουμε ότι τριπλασιάζουμε, τουλάχιστον τριπλασιάζουμε τον προπολογισμό για τη διαφήμιση, το οποίο είναι θετικό βεβαίως, αλλά πρέπει να επισημάνω και πάλι ότι δεν θα είμαστε σε θέση να τα κάνουμε όλα μόνο μέσα από τη διαφήμιση. Στο μέλλον θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα προϊόντα θα είναι προσβάσιμα στους καταναλωτές. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια εγώ. Λοιπόν, Τώρα αναπτύσσουμε αυτή την πολιτική για την ενημέρωση. Ένα είδος εξαγωγικής ε, επιδότησης, βοήθειας κλπ. Και πράγματι ε, προωθούμε τα μέτρα βιαστικά, σαν να καταπολεμούμε μια πανδημία. Εγώ τα φοβάμαι όλα αυτά τα θέματα τα οποία συζητούνται στο τέλος της θητείας για τα οποία θέματα δεν υπάρχει επαρκής χρόνος και το κάνει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας το κάνει. Ξέρω ότι χαμογελάτε σας βλέπω κύριοι όμως θέλω να παρουσιάσω και τη δική μου θέση από αυτού. Και κατευθυνόμεθα προς πιο κεντρική διαχείριση, ίσως να είναι αποτελεσματικότερη και ίσως να είναι ένα είδος παρέμβασης μέσω προώθησης προϊόντων. Όμως αυξάνουμε επίσης και τους πόρους. Αυτό είναι καλό. Αλλά περιορίζουμε την συγχρηματοδότηση προς όφελος οργανισμών, προς όφελός τους, κυρίως λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωργοί και κυρίως στα νέα κράτη-μέλη, οι δεν είναι καλά οργανωμένοι. Αυτές οι οργανώσεις εκεί των παραγωγών είναι ακόμα στην παιδική τους ηλικία, αν μπορώ να το πω έτσι. Εξού και ανησυχίε μου όσον αφορά όλα αυτά που συζητάμε Αυτές οι ανησυχίες πιστεύω πρέπει να ληφθούν υπόψη, διότι για την προώθηση, για την ενημέρωση, για τα προϊόντα είναι μια διάσταση πολύ σημαντική αυτή. Αυτές όμως είναι βάσιμες ανησυχίες που εκφράζω. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Γενικής Διευθύνσεως Γεωργίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε το λόγο. Και μετά ε, ο εισηγητής θα ξανά το λόγο. Η εισηγήτρια θα έχει ξανά το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω ε, που η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γνώρισε αυτή την υποδοχή για τις ενέργειες ενημέρωση σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα ε, είναι πολύ θετική. Τι στόχους έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, τα είπε ήδη ο Επίτροπος, ο Επίτροπος Τσόλος σε προηγούμενη συνεδρίαση. Αν θέλετε μπορείτε να τα βρείτε. Ε, ε, μπορεί να τα χαρακτηρίσει κανείς ότι πιάνουν περισσότερο τόπο τα χρήματα των φορολογουμένων. Απλούστευση, δικαιοσύνη και πιο εύκολη ελεξιμότητα. Είναι η λέξη κλειδιά εδώ. Επιτρέψτε μου τώρα να αναφερθώ σε κάποιες τροπολογίες, όχι όλες, για να εξηγήσω για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει διαφορετικό δρόμο σε πολλούς τομείς. Καταρχάς, ε, για την ενημέρωση και την προώθηση. θα πρέπει να είναι αυτή η ίδια για την εγχώρια αγορά, την εσωτερική και για τις τρίτες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της ε, προτείνει να χρηματοδοτείται η πρόθεση μόνο για τρίτες χώρες. Εάν θέλουμε και για την εσωτερική αγορά να τα χρηματοδοτούμε από τον κοινοτικό προπολογισμό, αυτό τι σημαίνει. Για παράδειγμα, η βελγική σοκολάτα που αναφέρθηκε, θα διαφημίζετε και θα προωθείτε και στο Βέλγιο. Και θα αναφέρει τη βελγική προέλευση και τα σήματα και θα ε, απευθύνονται στον ε, Βέλγο καταναλωτή. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προτείνει κάτι τέτοιο διότι πιστεύει ότι αυτό το ίδιο ευρώ που θα δαπανηθεί εκεί είναι, πιάνει περισσότερο τόπο εάν κάνουμε διαφήμιση σε τρίτες χώρες και όχι στην εσωτερική αγορά για την πρόθεση αυτών των προϊόντων. Εξού και η λογική. 75% των μέσων. Για τρίτες χώρες, χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό το ποσοστό. Στην εσωτερική αγορά η ανάλυση Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει ότι έχει νόημα να κάνουμε εκστατείες πληροφόρησης, όχι προώθησης. Αλλιώς θα υπάρξουν προβλήματα στρέβλωσης ανταγωνισμού. Στη συνέχεια, ποια προϊόντα θα καλύπτονται τώρα από αυτά ε, τα μέτρα και θα μπορούν να προωθούνται. Όλα που είναι στο παράρτημα 1, τα γεωργικά προϊόντα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να εξαιρεθεί το ψάρι, γιατί υπάρχει... Ε, για τα αλλιεύματα και τα προϊόντα ηχθείων άλλη ε, διαταξή σε άλλο κανονισμό και δεν θα πρέπει να έχουμε επικαλύψεις. Για το κρασί τώρα θα πρέπει να μην έχουμε ξεχωριστά εδώ στην κοινή οργάνωση αγορές για τα προϊόντα ίνου έχουμε 145 εκατομμύρια δεν μπορούμε να προωθούμε ξεχωριστά το κρασί. Αν θέλετε μαζί με άλλα προϊόντα, καλώς. Nicht ε, Προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όχι μόνο αυτά που αναφέρονται στο παράρτημα 1, αλλά και τρόφιμα τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα κατάλογο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο πριν από 1,5 περίπου χρόνο. Η τροποποίηση και η τροπολογία που προτείνεται θα μπορούσε ενδεχομένω να καλύπτει ε, και προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, αλλά είναι γεωργικά προϊόντα. Και είναι πάρα πολύ ασαφές. Θεωρητικά θα μπορούσαμε να προωθούμε ακόμα και δερμάτινα μπουφάν. Γιατί όχι, ζωικά προϊόντα. Είναι και το δέρμα μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι προϊόν της γεωργίας. Ε, όχι. Ε, και μόνο 20% της εκστρατείας να καλύπτει αυτό. Κατά τη δική μας ε, άποψη αυτό γνωρίζει πρακτικές δυσκολίες για τον έλεγχο του. Γιατί δεν είναι καθόλου σαφές πώς αυτό το 20% μπορεί να γίνει αντιληπτό περιορισμός και μετά ποιος και με ποιο τρόπο θα κληθεί να τα ελέγξει. Θεωρείται λοιπόν αυτό όχι απλούστευση αλλά ε, δυσχέρεια της πρότασης για την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη συνέχεια, ακούστηκε η δυνατότητα ενημέρωση σε περίοδους κρίσης ή καταστάσεις κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εσκεμένα δεν έχει προβλέψει τέτοια μέτρα βράχη πρόθεσμα σε περιπτώσεις κρίσεων, διότι από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο πριν από λίγο καιρό εγκρίθηκε ένα μέτρο ή μάλλον δύο μέτρα τα οποία καλύπτουν αυτή τη βραχή πρόθεσμη δράση. Το ένα είναι στην κοινή οργάνωση ε, αγοράς και το άλλο στην εγκάρσια, την οριζόντια. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει η εθνική συγχρηματοδότηση να καταργηθεί ως δυνατότητα. Για ποιο λόγο, για να υπάρχει ισότητα και δικαιοσύνη απέναντι σε όλους τους δεχόμενους αποδέκτες και δικαιούχους. Υπάρχουν κράτη-μέλη και περιφέρειες που δεν έχουν τα χρήματα για να κάνουν την εθνική συγχρηματοδότηση. Και για να μην αντικηθεί κανείς και να είναι όλοι στην ίδια κατάσταση ανταγωνισμού, πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακριβώς για λόγους δικαιοσύνης η εθνική συγχρηματοδότηση να καταργηθεί. 60% σε πολλές περιπτώσεις ζητά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν χρειάζεται αυτό για μικρομεσαίες να γίνει 75% ο συντελεστής το ποσοστό και πάλι υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες διότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κανονικά είναι ένα τμήμα ε, των οργανώσεων παραγωγών, έτσι δεν είναι. Οι οποίες οργανώσεις ε, είναι οι συνομιλητές και οι δικαιούχοι για μέτρα προώθησης ε, της εμπορίας των προϊόντων και πάλι ε, θα υπήρχαν μεγάλες δυσκολίες ελέγχου εάν πάμε στο 75% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, εμείς πώς κατανοούμε συλλογικά την πρόταση. 75% κοινοτική χρηματοδότηση συν 20% από εθνικά χρήματα θα μπορούσε για να φτάσουμε τελικά σε ένα ποσοστό της τάξης των 95% για προϊόντα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό σημαίνει υψηλότερη επιδότηση από ό,τι μέχρι τώρα. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταλήγει ε, στο γεγονός ότι δεν θα πρέπει να θίγεται η ευστοχία και αποτελεσματικότητα ε, και να εξασφαλίζεται από τους ίδιους τους παραγωγούς. Όταν έχουμε τόσο υψηλή ε, επιδότηση ε, να αυξάνεται επιπλέον. Υπάρχει κίνδυνος να αποβεί αυτό εις βάρος ποιότητος. Ένα άλλο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γίνεται μόνο μια προκήρυξη ετησίως. Αυτό συνάδει και με άλλα προγράμματα, όπου είναι τις οι διαγωνισμοί και οι προκηρύξεις τους. Γιατί είναι ετήσια και η στρατηγική που καθορίζεται κάθε φορά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι αυτό είναι πιο εύκολο και για τη διοίκηση, γιατί όταν είναι εξαμηνιά η προκήρυξη θα πρέπει όλα να τα ελέγχουμε δύο φορές το χρόνο. Εάν είναι μία φορά το χρόνο, όλα τα προγράμματα ε, που ξέρουν ποιοι είναι οι δικαιούχοι μπορούν να αξιολογούνται από κοινού και να επιλέγονται τα καλύτερα προγράμματα και για την ε, υλοποίηση αυτής της στρατηγικής. Και πάλι πιστεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έτσι έχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και υψηλότερη προστιθέμενη αξία για τα χρήματα των φορολογουμένων. Πιάνουν περισσότερο τόπο δηλαδή. Αυτές οι παρατηρήσεις είχε να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευνοϊκή υπόδοχη που επιφυλάξατε ουσιαστικά στην πρώτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον εκπρόσωπο της ε, Κομισιόν. Το, λόγο έχει η κεντρία. Ευχαριστώ κύριε Σικέρσκη, ευχαριστώ και τους συναδέλφους για τις τοποθετήσεις τους. Υπάρχει μια ισπανική παροιμία που λέει ε, να με ντύσετε αργά γιατί βιάζομαι. Μάλλον ντύνομαι αργά γιατί βιάζομαι. Που σημαίνει σπέβδε βραδέως. Καλά να κάνουμε τα πράγματα με ουσία και το θέμα δεν είναι να τρέχουμε άρον-άρον, να φτάσουμε πρώτοι και να έχουμε ένα κακό αποτέλεσμα. Τώρα είπατε ότι σας άρεσε το κείμενο. Ξέρετε ότι το έχω γράψει σε λιγότερο από 8 εβδομάδες και ήταν και κατά μεσής Χριστούγεννα. Δηλαδή μπορεί κανείς να δουλεύει υπό πίεση και με χρονική ε, ακριβώς τέτοια πίεση ε, κάνει κάποιες θυσίες από τον ελεύθερο χρόνο, από την ανάπαυση, από την αναψυχή χωρίς να είναι αυτό εις βάρος της ποιότητας. Αν μπορούμε γρήγορα να δουλεύουμε και ποιοτικά, ακόμα καλύτερα. Αυτό κάναμε. Ο κύριος Νίκολσον αναφέρθηκε σε ποσοστά. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε. Προς χώρες, πόσα και πόσα προς την εσωτερική αγορά. Όπως σας είπα προηγουμένως, εγώ δεν έχω κάνει πρόταση για το πώς θα κατανεμηθούν αυτά τα κονδύλια να περιμένουμε να δούμε τι θα προτείνουν οι συνάδελφοι, πώς το βλέπουν οι πολιτικές ομάδες, πού πρέπει να κινηθεί αυτό το ποσοστό, πόσο μέσα, πόσο έξω και τελικά να συμφωνήσουμε, αν γίνεται, ε, με συμβιβασμούς για να έχουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη συμφωνία για τις προτάσεις αυτές. Πόσο θα απευθύνεται στην εσωτερική αγορά και πόσο για τις τρίτες χώρες. Είναι γεγονός, ακούστηκε προηγουμένως, ότι η ουσιαστική αγορά είναι εσωτερική μας, αλλά επίσης το δυναμικό αύξησης είναι στις τρίτες χώρες. Περιμένω λοιπόν τις τροπολογίες των συναδέλφων. Δηλαδή, όσο περισσότερο συμφωνούμε, τόσο καλύτερο. Κάποιος ρώτησε, ο συνάδελφος Ρούμπιξ, που έχει φύγει τώρα, ποιος είναι ο στόχος μας. Ο στόχος μας είναι να πουλάμε τα προϊόντα μας και εντός και εκτός της Ένωσης. Η γεωργία, η κτηνοτροφία και ε, η βιομηχανία τροφίμων αυτό που θέλει είναι να πουλάει. Και γι' αυτό χρειάζεται αυτό το μέσον. Θα πρέπει να κοιτάμε συλλογικά τις πωλήσει για τον κλάδο χωρίς να έχουμε μονές σε συγκεκριμένους στόχους ενιαίους για όλους, ένα κορσέ. Εμεί ενδιαφερόμαστε να πουλάμε και στι τρίτε χώρε και στους καταναλωτές τους, να γίνουν γνωστά τα προϊόντα μας, ε, όπως και στους ίδιους του Ευρωπαίους πολίτες. Ε, θυμάστε ότι υπήρχε μια στρατηγική για την ποιότητα με εισηγήτρια την κυρία Γκαρσία Πέρες και λέγαμε και συμφωνήσαμε όλοι ότι θα πρέπει οι πολίτες να γνωρίζουν τις δικές μας ποιοτικέ μάρκες που ήταν πολλές, πολύ αξιόλογες και ποιοτικέ και ο κόσμος δεν τις γνώριζε. Στόχος λοιπόν είναι οι πωλήσει εντός και εκτός της ενώσεως. Γι' αυτό λέγω ότι είναι για μένα το σημαντικότερο. Είπε ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής δύο προκήρυξεις το χρόνο, μία προκήρυξη διαγωνισμού το χρόνο. Εμείς γιατί επιμένουμε για τις δύο. Μα όταν έχεις στρατηγική, και συγκεκριμένους στόχους για μια τριετία. Γιατί έτσι δουλεύει το μάρκετινγκ και η διαφήμιση. Εκείνος λέει μια φορά το χρόνο προκηρύξεις γιατί είναι πιο εύκολο για εκείνους. Ο κλάδος ζητάει δύο φορές το χρόνο. Τώρα τι θα κάνουμε. Είναι περισσότερο διαδικαστικό αυτό το θέμα παρά ουσιαστικό η πολιτική θέση. Τι λειτουργεί καλύτερα και τι είναι πιο λογικό. Εκεί θα πρέπει να συμφωνήσουμε, μάλλον σε τεχνική βάση περισσότερο και λιγότερο πολιτική. Γιατί πολιτικά τι μας ενδιαφέρει, επαναλαμβάνω, να αυξηθούν οι πωλήσει των προϊόντων μας. Λέτε ότι υπάρχουν αρκετά λεφτά στην κοινή οργάνωση αγοράς για τον ίνο και για τα άλλα προϊόντα. Λυπάμαι να διαφωνώ και να αντιλέγω με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν ήταν αρκετά τα κονδύλια και αρκετές ε, οι θέσεις, δεν θα είχαμε ζήσει το σκάνδαλο με την Σερίχια Κόλλη στον βαθμό αυτό. Και αν είχαν πάρει εγκαίρος ε, όπως έπρεπε, τη βοήθεια, ε, μάλλον θα είχαν πάρει εγκαίρος και όπως έπρεπε τη βοήθεια τους η παραγωγή. Λυπάμαι που διαφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Κοινοβούλιο, αλλά θα πρέπει να το σκεφτεί λίγο παραπάνω αυτό. Διότι πρώτον, τους δίνουμε τη δυνατότητα άμεσης αντίδρασης ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περισσότερη εξουσία να αντιμετωπίσουν προβλήματα και επίσης πιστεύω ότι είναι σημαντικό αυτό το εργαλείο για αυτές τις κρίσεις που ξεσπάνε στην αγορά. Τώρα, για τα μέσα ποιότητας δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με αυτό το κείμενο είναι να πουλήσουμε ευρωπαϊκή εικόνα, ευρωπαϊκή ποιότητα και ευρωπαϊκές προδιαγραφές παγκοσμίω εντός και εκτός της ενώσεως. Και επειδή υπάρχουν ήδη εθνικά προγράμματα, αρκετά επαρκή, που μπορούν να προωθούν τα ντόπια σήματα που δεν έχουν πανευρωπαϊκή εμβέλεια, ας ασχοληθούμε με τα ποιοτικά προϊόντα που έχουν πανευρωπαϊκή εμβέλεια, χωρίς αυτό να υποτιμά καθόλου ε, τα τοπικά προϊόντα, τα οποία όμως πολλούνται στην εγχώρια αγορά και έχουν τα απαραίτητα εργαλεία προώθησης και διαφήμισης. Αυτά. Ελπίζω να μην ξέχασα τίποτα. Σας ευχαριστώ όλους για τις παρεμβάσεις και για την υποστήριξή σας. Περιμένω τις τροπολογίες σας και από τις 14 του μηνός και μετά θα συμφωνήσουμε όσο γίνεται περισσότερο έτσι ώστε να μπορέσουμε με όλες τις δυνάμει να πάμε να διαπραγματευτούμε με Συμβούλιο και Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Συγήτρια. Όπως είπατε, η προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι η 14η Φεβρουαρίου, η μερα Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι. Και θα εξετάσουμε την έκθεση αυτή στις 18 Μαρτίου και τον Απρίλιο θα περάσει την Ολομέλεια. Νομίζω ότι μπορούμε να μείνουμε εδώ. Σας ευχαριστώ όλους. Ε, θα επανέλθουμε αύριο το πρωί στις 9. Καταφέραμε να ολοκληρώσουμε και 15 λεπτά νωρίτερα. Γεια σας.